Colleagues. Ε, συνάδελφοι καλημέρα. Παρακαλώ να καθίσετε. Και παρακαλώ από τους δημοσιογράφους να βγουν από την αίθουσα. Θέλω να καλωσορίσω στη συνεδρίαση της ε, Οικονομικής Επιτροπής τους Υπουργούς κυρίως κυρίους Σόιμπλε και Παντοάν. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μας και τιμή μας να έχουμε μια συζήτηση με δύο από τους πιο επιφανείς Υπουργούς Οικονομικών σημαντικούς όχι μόνο σε σχέση με το ΑΕΠ που εκπροσωπούν, αλλά και σε σχέση με τις θέσεις τις οποίες έχουν εκφράσει σε τομείς καθοριστικούς για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Δεν ταυτίζονται οι απόψεις τους, αλλά ταυτίζονται σε σχέση με την αντίληψη που έχουν και την ανάγκη να υπάρξουν περαιτέρω βήματα για μια πιο ολοκληρωμένη και δημοκρατική οικονομική και νομισματική ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα στα πλαίσια της έκθεσής μας για την οικονομική διακυβέρνηση. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Μπερές. Η ανταλλαγή αυτή απόψεων γίνεται και στα πλαίσια μιας ενδιαφέρουσα συγκυρίας. Το θέμα της ευελιξίας που θεωρούμε ότι θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε σωστά κάποια από τα χαρακτηριστικά του Συμφώνου για την Ανάπτυξη, κάποια νέα χαρακτηριστικά επίσης της νέας οικονομικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επίσης ε, και τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα είναι όλα θέματα που θα καταστήσουν ε, τη συζήτησή μας ιδιαίτερως ζωηρή. Η πρώτη εισαγωγική παρατήρηση θα γίνει από τον κύριο Παντοάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Αγαπητέ Βολφκανγκ. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που έχω την δυνατότητα να ανταλλάξω απόψεις με σε ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο η οικονομική διακυβέρνηση της ε, ε, Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Η αξιολόγηση του πλαισίου του ισχύοντος ε, θα πρέπει να βασίζεται το σε ποιο τρόπο η διακυβέρνηση μέχρι τώρα έχει οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της περαιτέρω ολοκλήρωσης και μιας ανάπτυξης πλούσιας σε απασχόληση και ισόρροπης και σε μια φυσικά πορεία οικονομικής σύγκλησης, υψηλότερης σύγκλησης. Νομίζω ότι ο απολογισμός δεν είναι ικανοποιητικός και γι' αυτό εδώ θα σταθώ έτσι ώστε να δούμε τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από την εμπειρία που σωρέψαμε μέχρι τώρα για το μέλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ σε πέντε σημεία, τα οποία νομίζω με συνθετικό τρόπο παρουσιάζουν τα συμπεράσματα της εμπειρίας την οποία βιώσαμε όλοι. Το πρώτο είναι ότι μια αποτελεσματική διακυβέρνηση θα πρέπει να βαθίζεται σε ένα συνεκτικό policy mix, σε ένα συνεκτικό μείγμα πολιτικής και σε επίπεδο δημοσιονομικό και σε επίπεδο διαρθρωτικό και σε επίπεδο χρηματοπιστωτικό και φυσικά σε επίπεδο ε, νομισματικής, οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Πρέπει να υπάρχει ένα σωστό συντονισμός αυτών όλων έτσι ώστε να υπάρξουν θετικά βήματα. Η διαπίστωση αυτή γεννιέται και από μία άλλη διαπίστωση και θα είμαι πολύ συνεκτικός εδώ για την κρίση η οποία οδήγησε εδώ και λίγα χρόνια σε μια ευαίσθητη θα έλεγα κατάσταση το ευρώ. Η κρίση του ευρώ έδειξε ότι στα πλαίσια μιας οικονομικής ένωσης μπορεί να αναπτυχθούν ανισότητες, ανισορροπίες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στα πλαίσια της σχεδίασης της αρχιτεκτονικής της. Τέτοιου είδους ανισορροπίες μπορεί να ε, καταστούν πολύ επικίνδυνες. Απαιτείται να χρησιμοποιηθούν με συντονισμένο τρόπο όλα τα διαθέσιμα μέσα. Και αυτό με τη σειρά του ε, επιζητεί και επιβάλλει μια ενίσχυση της ε, governance, της διακυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να καλύπτονται οι ανισότητες αυτές σε σωστό χρόνο και κυρίως να προλαμβάνονται έτσι ώστε να μην καταστούν ε, μη αντιμετωπίσιμες πλέον και ε, οδηγήσουν σε ε, πολύ σημαντικότατα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν η δομή της διακυβέρνησης και μπορούμε να το πούμε εύκολα αυτό το συμπέρασμα να είναι πιο αποτελεσματική. Έγιναν πολλά και σε επίπεδο συντονισμού και σε σχέση με την παρουσίαση σαν παράδειγμα των εθνικών προϋπολογισμών στο Eurogroup. Αλλά πολλά μένει να γίνουν για τον καθορισμό μιας συνεκτικής στρατηγικής η οποία να εξετάζει με συστηματικό τρόπο τον υπερεθνικό χαρακτήρα των συνεπειών της πολιτικής της κάθε χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο οι εθνικές πολιτικές και η ευρωπαϊκή πολιτική μεταξύ τους λειτουργούν διαδραστικά αυτό με οδηγεί στο δεύτερο συμπέρασμα από την πορεία μας μέχρι τώρα, το λεγόμενο spill over, οι επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής μιας χώρας στις άλλες χώρες. Αυτά τα spill over, αυτές οι επιμολύνσεις μπορεί να αναλυθούν, να εξεταστούν με πιο προσεκτικό τρόπο στις αποφάσεις για την μελλοντική πολιτική, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν μια αποτελεσματική αξιολόγηση των λεγόμενων spill over όπως ε, λέει και η διεθνής εμπειρία να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και να βελτιώσει τις επιδόσεις ε, της ε, οικονομικής περιοχής, του οικονομικού χώρου του οποίου την οικονομική διακυβέρνηση θέλουμε να ενισχύσουμε. συγκεντρώσαμε μέχρι τώρα την προσοχή μας στις αρνητικές μορφές ε, ε, επέκτασης, αν θέλετε, κάποιων αρνητικών στοιχείων των εθνικών πολιτικών. Στο μέλλον η διακυβέρνηση προφανώς και θα ελέγχει και τις αρνητικές πλευρές, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει και στην αξιολόγηση των θετικών πλευρών. Ένα τρίτο σημείο είναι να πούμε ότι απαιτείται μια καλύτερη και επακριβέστερη συμπληρωματικότητα των εθνικών πολιτικών με την ευρωπαϊκή πολιτική. Οι μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές σε επίπεδο εθνικό που είναι αν θέλετε το κομβικό σημείο μιας ουσιαστικής οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο συνεκτικό με ευρωπαϊκό όραμα, με ευρωπαϊκή στρατηγική ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα εθνικά μέτρα και τα κοινοτικά μέτρα να συνδυάζονται και αναφέρομαι εδώ στην πλήρη εφαρμογή της ενιαίας αγοράς. Η ενιαία αγορά είναι καταπληκτικός μηχανισμός ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο η απλούστευση των ε, φορολογικών συστημάτων όπως επίσης και μια πραγματική ένωση της αγοράς κεφαλαίων, το Capital Markets Union. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να διασφαλίσουν μια περαιτέρω συνεκτικότητα και θα πρέπει να φαίνονται και στα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε την κατάσταση όπως η ετήσια ε, ε, ε, έκθεση για την ανάπτυξη. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο συγκυριακό. Οι δράσεις της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα της διαφορετικής αυτής πλευράς, ε, επηρεάζουν ε, με, θα έλεγα, σε μια πολιετή προοπτική τα πράγματα. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ένα σωστός χρονισμός στην σύλληψη, τη σχεδίαση και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, όπως και τον υπολογισμό των επιπτώσεων που έχουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές στα πλαίσια των οικονομικών πολιτικών. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε ακόμα περισσότερο, να αξιολογούμε δηλαδή με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις προσπάθειες τις οποίες κάθε χώρα οφείλει να προωθήσει στα πλαίσια της εθνικής οικονομικής της πολιτικής. Αυτό θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η διαρθρωτική διάσταση και η μακροοικονομική διάσταση των πολιτικών που ακολουθούν οι διάφορες χώρες ε, ε, μεταξύ τους αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι θα βελτιστοποιήσουμε την δράση της ε, οικονομικής μας πολιτικής μέσα στον χρόνο και σε εθνικό επίπεδο και σε κοινοτικό επίπεδο. Ένα τελευταίο σημείο. Ίσως αυτό να είναι και το πιο σημαντικό, ίσως. Είναι η ανάγκη να ενισχύσουμε και την εθνική ευθύνη, την αίσθηση ιδιοκτησίας των οικονομικών προγραμμάτων, το ownership των οικονομικών πολιτικών, αλλά και να προωθήσουμε επίσης και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εγώ προσωπικά πιστεύω κάποια, ότι κάποια μέτρα οικονομικά, κάποια μέτρα οικονομικής πολιτικής που έχουν σωστά παρουσιαστεί και έχουν σωστά εφαρμοστεί, ε, παρουσιάζουν κάποια αποτελέσματα κατώτερα, κατώτερα των ε, αναμενόμενων ε, Τώρα μου είπαν ότι το ρολόι που έχω μπροστά μου δεν δείχνει τον σωστό χρόνο. Υπάρχει ένα θέμα με το χρόνο. Και διακόπτει ο κύριος Παντών. Λοιπόν, το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης τίθεται εδώ. Πολλές δράσεις της οικονομικής πολιτικής σχεδιάζονται σωστά, εφαρμόζονται σωστά και παράγουν καρπούς κατώτερους μερικές φορές των προσδοκιών γιατί δεν είναι σε θέση να προκαλέσουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη και ενδιαφέρον ε, στους εμπλεκομένους. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της πολιτικής όμως, να προσπαθήσουμε να παρουσιάζουμε τα μέτρα αυτά με σωστό και κατανοητό τρόπο, με ευκρινή τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξει μια ένεση εμπιστοσύνης ε, μέσω των οικονομικών αυτών πολιτικών. Αυτό ισχύει, επαναλαμβάνω, και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ υπάρχει ένα τελευταίο σημείο, δηλαδή ο καθορισμός του πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης δεν θα πρέπει να αποκρύβει τη σημασία που έχουν οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορεί και να μην έχουν άμεσες, ε, όσοι πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική πολιτική, είναι λάθος γιατί υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο που αυξάνουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και επηρεάζουν με καθημερινό τρόπο την ζωή των πολιτών μας και την οικονομική κατάσταση σε πολιετή βάση. Και έτσι μεγιστοποιούν αν θέλετε και τις οικονομικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, η θεσμική διακυβέρνηση από τη μία και η οικονομική από την άλλη πρέπει να συνδυάζονται. Ευχαριστώ κύριε Πάντο. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό Σόιμπλε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ενώπιον της Επιτροπής σας. Ο Κάρλο Παντοάν προείδρευε στο ΕΚΟΦΗΝ. Ήταν ο πρόεδρός μου πριν από μερικές εβδομάδες. Πολύ καλός πρόεδρος. Και γι' αυτό και του άφησα και λίγο από το χρόνο της ομιλίας μου. Θα κάνω μόνο μερικές σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα δίνει την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ξεκινήσει από την καλή πλευρά τη ζωή του και βρίσκεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Δεμπρόφσκης, εχθές στην Επιτροπή, έκανε μια πολύ βασική νομίζω παρατήρηση και είπε ότι το risk sharing και το sharing of sovereignty, δηλαδή ο επιμερισμός του κινδύνου και ο επιμερισμός της κυριαρχίας, πάνε χέρι-χέρι. Άρα Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, για όλους αυτούς τους καλούς λόγους που περιέγραψε ο κύριος Παντοάρ μόλις τώρα, χρειάζονται αλλαγές στο πρω... πρωτογενές δίκαιο, στο νομικό πλαίσιο. Γιατί ακριβώς στο νομικό αυτό πλαίσιο, του πρωτογενές δίκαιο, έχουμε ένα θεσμικό πρόβλημα. Πρέπει να τροποποιηθεί λοιπόν αυτό, όπως ζητεί πάντα η κυβέρνηση της Γερμανίας και στο βαθμό που δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε, δεν έχουμε μπορέσει ακόμη να τροποποιήσουμε το πρωτογενές δικαίωμα, θα πρέπει με το ισχύον πλαίσιο, μέσα στο ισχύον δηλαδή πλαίσιο των συνθαϊκών, να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και συνεργασία μέσα στην Ευρωζώνη για όλους αυτούς τους λόγους που είναι ήδη γνωστοί και που ήδη ο Κάρλο ανέφερε. Καθοριστικό πάντως είναι οι κανόνες στους οποίους έχουμε καταλήξει, στους οποίους έχουμε συμφωνήσει να τηρούνται. Αυτό είναι το βασικό γιατί έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κυρίως της Ευρωζώνης. Ότι δηλαδή οι συμφωνίες, οι κανόνες που εμείς οι ορίζουμε τηρούνται. Άρα, οποιαδήποτε σκέψη για ε, πιο ελαστική εφαρμογή των κανόνων πλήττει όχι μόνο τους ίδιους τους κανόνες, αλλά και την εμπιστοσύνη για τα υπεσχημένα, για τα συμπεφωνηθέντα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά από την ίδρυση της Ευρωζώνης, γιατί εγώ τότε ήμουν ήδη παρόν και δραστήριο στα πολιτικά, Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι η ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη Δημοσιονομική και Οικονομική Ένωση ήταν ανέκαθεν το κύριο διαφιλονικούμενο ζήτημα. Και πάντοτε συζητούσαμε αν μπορούμε να καταφέρουμε μια νομισματική ένωση χωρίς τη Δημοσιονομική και Οικονομική Ένωση και επίσης εκφραζόταν το αίτημα ότι θα χρειαστεί μια ε, διακυβέρνηση. Ή αν θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε πρώτα την πολιτική ένωση, πράγμα το οποίο ίσω ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, ή αν θα έπρεπε να προχωρήσουμε προς κάποιου πιο ε, κανόνες πιο σαφή. Οι οποίοι δεν έχουν τηρηθεί πάντα όμω. Και εγώ προέρχομαι από κράτο το οποίο δεν έχει τηρήσει του κανόνε από την αρχή και πολλοί εταίροι μα δεν το έχουν λησμονήσει αυτό. Εμεί όμω τα αποκομίσαμε τα διδάγματα αυτά. Όταν ε, την εποχή εκείνη αναλάμβανε καθήκοντα η καγκελάριο στη Γερμανία, είχε χρειαστεί να εξηγήσει με τον Υπουργό των Οικονομικών Στάινμπρουκ την εποχή εκείνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη και ότι δεν πρέπει να ε, προχωρήσουμε με τον τρόπο αυτόν και ότι υπάρχει ζήτημα ελλείμματος της Γερμανίας. Αυτό το λόγο ακριβώς θέλουμε εμείς να τηρούνται οι κανόνες γιατί έχουμε αποκομίσει τα διδάγματα. Και έχουμε αποκομίσει επίσης και τα διδάγματα της αλληλεγγύης η, ευρωπαϊκή, η οικονομική κρίση, η τραπεζική κρίση μας έδειξε ότι πολύ γρήγορα μπορούν οι χρηματοπιστωτικές χώρες να χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε ένα οικονομικό σύστημα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει και στο θέμα αυτό να στραφούμε, έστω και αν δεν έχουμε πάντα την καλύτερη λύση. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα περίπλοκο πλαίσιο ρύθμισης που στόχο είχε την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ε, Ευρωζώνη με ανάληψη και εκδήλωση σημαντικού βαθμού αλληλεγγύης για πολλά κράτη της Ευρωζώνης, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, αλλά μην το λησμονούμε. Δεν υποχρεώσαμε κανένα να λάβει καμία δέσμευση. Δείξαμε τεράστια αλληλεγγύη και ήμασταν διατεθειμένοι να τη δείξουμε διότι θεωρήσαμε ότι καθιστούσε απαραίτητη την εκδήλωση της ελληνικής στο κοινό συμφέρον όλων των Ευρωπαίων. Αλλά η αρχή που είναι γνωστή και από την αναπτυξιακή πολιτική και εγώ τη γνωρίζω γιατί η γυναίκα μου δούλευε πολλά χρόνια στην αναπτυξιακή πολιτική που λέει σε βοηθώ για να μπορείς να βοηθηθείς σημαίνει ότι πρέπει να επιληθούν τα βασικά προβλήματα και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Να λαμβάνονται στα κράτη-μέλη οι ορθές εκείνες αποφάσεις οι οποίες θα επιτρέπουν στην Ευρώπη να αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα τις μεγάλες αυτές προκλήσεις που τόσο γρήγορα μπορεί να εμφανίσει η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και που μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη πρόκληση για η αδίποτε ευρωπαϊκή οικονομία εφόσον δεν μπορεί να έχει ένα γερό κοινωνικό σύστημα, ένα σύστημα απόδοση, παραγωγικής οικονομίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε συνηθισμένοι σε ένα πολύ καλό κοινωνικό σύστημα και σε ένα ε, ε, σταθερό παραγωγικό σύστημα, πολύ περισσότερο από ό,τι άλλα κράτη, αλλά θα πρέπει αυτό να το λύσουμε, να το δούμε σε ένα ζήτημα όχι δογματικό, αλλά σε ένα ζήτημα ανάγκης και εξυπηρέτηση της λειτουργία των δημοκρατιών και των οικονομιών μας. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε με την επεξεργασία αυτής της μεταρρύθμισης Ευρωζώνης, γιατί νομίζω ότι προχωρήσαμε αρκετά την προηγούμενη χρονιά με σταθεροποίηση του ευρώ, με παροχή βοήθεια στα κράτη τα οποία είχαν ανάγκη και δεν μπορούσαν να πωλήσουν ομόλογα στις διεθνείς αγορές, τους προσφέραμε μεγάλη βοήθεια και πάντοτε λέγαμε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι ρίζες τα αίτια των προβλημάτων. γιατί δεν έπρεπε να δοθεί εσφαλμένη εντύπωση ε, που δόθηκε ορισμένες φορές σε ορισμένα κράτη ότι κάποιος άλλος θέλει. Τα προβλήματα ξεκινάνε πάντα στο εσωτερικό μιας χώρας και προσπαθούμε με αλληλεγγύη να βοηθήσουμε να λυθούν. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να τα λύσουμε στη θέση κάποιου άλλου. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σόιμπλε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, μετά στους σκιώδεις εισηγητές. Δύο λεπτά έχετε για τις ερωτήσεις και δυόμιση λεπτά για τις απαντήσεις και από τους δύο καλεσμένους μας. Οπότε δεν θα έχουμε 7 λεπτό όπως συνήθως. Μην υπερβαίνετε λοιπόν το δίλεπτο για την υποβολή των ερωτήσεών σας. Η κυρία Περβάς Μπερές, η συγγητριά μας. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το προνόμιο της συγγήτριας, ε, το δίλεπτο ολόκληρο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και τηλεγραφικά θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις μέσα στο δίλεπτο. Κύριε Πάντων, είπατε ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε τις ανισορροπίες για για να αποκτήσουμε μια ευρωπαϊκή επισκόπηση και θεώρηση των διακυβευμάτων. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε την αναθεώρηση του δίπτυχου και του εξάπτυχου πακέτου, γιατί αυτό, αυτή ήταν η βούληση του νομοθέτη. Είναι μια πόρτα που έχουμε ανοιχτεί μπροστά μας. Πιστεύετε ότι θα πρέπει αυτό να συνδυαστεί και με την ε, ανοιχτή συζήτηση για, τη, για την έκθεση των τεσσάρων προέδρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εθνικό επίπεδο και το ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, Έχετε κάποιε προτάσει, κάποιε ιδέε για να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο και η αποτελεσματικότητα του ισχύοντο μηχανισμού. Κύριε Σόιμπλε, επιμείνατε στην ανάγκη της στήριξη των κανόνων. Και το συμπέρασμά σα είναι ήταν ότι συνήθω το πρόβλημα προέρχεται από το εθνικό επίπεδο. Πόσο η εθνική κατάσταση αυτή εξηγεί την, την ύπαρξη όλο και μεγαλύτερων διαφορών στην Ευρωζώνη που υπήρχαν και πριν την κρίση αλλά επιδεινώθηκαν μετά την έξαρση της κρίσης και τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτές τις διαφορές και αποκλήσεις. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ε, δύσκολες και απαιτητικές. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπα προηγουμένως. Για το πώς θα βελτιώσουμε το δίπτυχο και το εξάπτυχο πακέτο και να χρησιμοποιήσουμε το όραμα των τεσσάρων προέδρων ε, ως κινητήριο δύναμη. Εν συντομία, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά από τον αντίκτυπο των μέτρων και την βιωσιμότητα του συστήματος, αν αναγνωρίσουμε πλήρως δύο πτυχές που προανέφερα. Τα διάφορα ε, μέσα και όργανα πολιτικής θα πρέπει να ενταχθούμε σε πιο ολοκληρωμένη διαδικασία. Για παράδειγμα, ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για ε, δεδομένη νομοθεσία και δεδομένη εφαρμογή ε, είναι διαφορετικός αυτός ο αντίκτυπος ανάλογα με το μακροοικονομικό κλίμα και περιβάλλον και τις εξελίξεις αυτού του μακροοικονομικού κλίμα, κλίματος. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ πολύ σωστά είπε ότι η νομισματική πολιτική έχει κάποιες δυνατότητες μέχρι ενός βαθμού, αλλά χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να αξιοποιηθούν πλήρως τα ωφέλη ενός καλού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Και ισχύει και το αντίστροφο οι διαστρωτικές μεταρρυθμίσεις θα λειτουργήσουν καλύτερα αν για παράδειγμα οι προβλέψεις ε, εξέλιξη των τιμών είναι σε ισορροπία και δεν έχουν μια φθήνουσα τάση όπως σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το όραμα των τεσσάρων προέδρων, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το όραμα για να διευρυνθεί ο ρόλος του συστήματος. Γιατί μπαίνουμε σε μια φάση όπου διάφορες χώρες βρίσκονται σε διαφορετική θέση σε ό,τι αφορά την πορεία προσαρμογής τους. Άλλες έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο, ε, ενώ μερικές υστερούν. Ε, αυτό όμως εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων. Αυτές θα πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει όμως και μια συστημική διάσταση που θα πρέπει να συμπεριληφθεί πιο ρητά και κατηγορηματικά από ό,τι στο παρελθόν δηλαδή να αναγνωριστούν ε, οι θετικέ και αρνητικές μεταδόσεις του αντικτύπου. Και βέβαια αυτά είναι κάπως γενικά σχόλια, αλλά μέσα σε μισή λεπτά αυτά πρόλαβα να πω. Ε, κύριε Σόιμπλε, κύριε Μπέρες, με ρωτήσατε το πώς εξηγώ το γεγονός ότι και πριν από την κρίση η εξέλιξη ορισμένων κρατών μελών μέσα στην Ευρωζώνη αλλά και της ίδιας Ευρωζώνης ήταν διαφορετική και άνεση. Καταρχάς δεν αποκλείεται μέσα σε ένα σύστημα ανταγωνισμού να υπάρχει σε αυτή τη συνύπαρξη ω συνέπεια του ανταγωνιστικού αυτού συστήματος διαφορετικά αποτελέσματα, ε, διαφορετικές επιδόσεις. Αλλά χρειάζεται βεβαίως συστήματα ισοστάθμισης. Ε, εξισωτικά συστήματα κατά κάποιο τρόπο. Όταν δηλαδή έχουμε να κάνουμε διαφορετικές κατάστασεις, να βρίσκουμε και διαφορετικές αναλογικές λύσεις. Αυτό είναι άλλωστε και το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εφαρμόζεται πάντοτε, όπως εφαρμόζεται άλλωστε σε κάθε ομόσπονδη, ομοσπονδιακή δομή. Εμείς από τη Γερμανία ξέρετε ότι έχουμε μακρά ομοσπονδιακή παράδοση. Μετά την ε, μετά το τέλος του δεύτερου της ε, ε, διχοτόμησης Γερμανίας που ακολούθησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου είχαμε πολλά υψηλά ποσά εκατομμύρια μάρκων που μεταφέρθηκαν οικονομικά στην Ανατολική Γερμανία από τη Δυτική για να στηρίξουν τις λιγότερο αποδοτικές οικονομίες της Ανατολικής Γερμανίας με χρήματα των πιο αποδοτικών εκείνων ε, κρατηδίων της Δυτικής Γερμανίας. Αυτό ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως θα πρέπει πάντοτε να γίνεται, όπως είπα, στο πλαίσιο των ισχύουσών συνθήκων και με βάση αμοιβαίας αλληλεγγύης. Αυτή η βάση της αμοιβαίας αλληλεγγύης είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή και να προσπαθούμε πάντοτε να τηρούμε τις συμβάσεις, τα συμπεφωνημένα, τους κανόνες. Βεβαίως νομίζω ότι από κοινού μπορούμε να επιλύουμε καλύτερα τα προβλήματα. Και βεβαίως θα πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στο εσωτερικό της Ευρώπης, αλλά να στρεφόμαστε και προς τα έξω και να βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση έξω από την Ευρώπη. Αυτό είναι γενικά το πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να μην επιβάλλουμε υπερβολικούς κανόνες σε βαθμό που να καταπνίγεται η λειτουργία μιας οικονομίας. Αυτό το λέω πάντοτε και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να καταπνίγεται, δεν πρέπει να συμπιέζεται η δυνατότητα η παραγωγική, η δυνατότητα, η δημιουργική μιας οικονομίας με την επιβολή υπερβολικά αυστηρών όρων το ίδιο το έχουμε δει εμείς στη Γερμανία και επιμένουμε. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με την ε, προόδο εφερειπίν που θέλουμε να επιδιώξουμε στη ψηφιακή οικονομία θα χρειαστούμε οπωσδήποτε απορρίθμιση για να έχουμε καλύτερο δυναμικό ανάπτυξης, μεγαλύτερο περιθώριο για επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Και θα πρέπει πάνω σε αυτό κυρίως, στην ψηφιακή οικονομία δηλαδή, να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ. Τώρα ο Σκιώδη ηγητής από το ΕΛΚ, η κυρία Έστερ Ντελάνκε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους δύο υπουργού που ήρθαν. Με ιδιαίτερη χαρά είδα το παρακαθήμενο του κυρίου Σόιμπλε να ανέβει ε, ε, συγκαταβατικά λέγοντα ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να το δούμε και με μια πιο παγκόσμια, παγκόσμια προοπτική. Μιλήσατε για την εμπιστοσύνη και οι δύο υπουργοί. Ωραία όλα αυτά αλλά τα συμπεράσματά σα ήταν κάπως διαφορετικά. Ο ένας μίλησε για, με, για... Ο είπε ότι η μεγαλύτερη ευελιξία θα οδηγήσει σε περισσότερη εμπιστοσύνη και ο άλλο είπε προσοχή με την ευελιξία μήπως επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Σόιμπλε. Τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα για περισσότερη ευελιξία ή είστε επιφυλακτικό. και προσεκτικό στο σημείο αυτό. Δεύτερο, μιλήστε για τι απαρχέ τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση και είπατε ότι δημιουργήσαμε την Νομισματική Ένωση αλλά δεν τηρήσαμε του κανόνε 2003, 2004 και το καθεξής. Πόσο επιζήμιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας να μην τηρήσουμε ούτε τώρα τους κανόνες που δημιουργήσαμε τις ημέρες της κρίσης. Πόσο επιζήμιο θα ήταν να τους παραβιάσουμε γιατί δεν του έχουμε αλλάξει. Κύριε Πάντο, μιλήσατε για το συμπατριώτη τον κύριο Ντράγκη, που πολύ σωστά είπατε ότι έχει τα όρια τη ε, η νομισματική πολιτική. Χρειαζόμαστε και διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Τώρα, να επικεντρωθώ στι μεταρρυθμίσει τη αγορά εργασία. Πόσο σημαντικέ είναι κατά τη γνώμη σα αυτέ σε μερικέ χώρε, όπω και στη δική σα πατρίδα, ε, ποιε πιστεύετε ότι θα είναι οι εξελίξει και τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Ελπίζω να μην ζητάτε δεύτερη ανακοίνωση για ευελιξία πολύ σημαντικό κάποιος τόσο έμπειρος ε, να μπορεί να μου πει τη γνώμη του γιατί το τι σημασία θα έχει κάτι τέτοιο για το μέλλον η ευελιξία αυτή. Πρώτα κύριε Σόιμπλε. Στην αρχή της τοποθέτησής μου έκανα την παρατήρηση ότι, στο πλαίσιο, ότι πρέπει να τηρήσουμε το νομικό πλαίσιο που ισχύει. Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι κακό η ευελιξία, αλλά δεν μπορεί η ευελιξία να υπονομεύει την εμπιστοσύνη. Και αν η ευελιξία οδηγεί στο να μην τηρούνται κανόνες στους οποίους έχουμε συμφωνήσει, και το είδαμε αυτό το 2003, τότε είναι λάθος ευελιξία, υπονομεύει την εμπιστοσύνη και έχει σημασία και πολιτική. Έχω μια σειρά λοιπόν από κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ σοβαρού πολιτικού που είναι πεπισμένοι για την ανάγκη τήρηση των καρόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πεπισμένο εδώ και δεκαετία. ότι οι πολίτε στα κράτη αυτά θέλουν να έχουν μία πρόοδο σταθερή και με ε, στόχο την Ένωση προς την, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το στόχο δεν τον έχουν εγκαταλείψει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παραμείνουν πιστές και οι διοικήσεις, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών με τον ίδιο τρόπο σε αυτούς τους στόχους. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντοτε. Στη Γερμανία και, και στη Γερμανία μπορούμε να μην τηρούνται πάντα οι κανόνες, αλλά δυστυχώς το βλέπουμε και σε άλλα κράτη-μέλη. Ελπίζω όμως να μην υπάρξει ένα πρόβλημα. Συγκεκριμένα παραδείγματα δεν θέλω να δώσω. Η εμπιστοσύνη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για, την, για τις οικονομικές επιδόσεις και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό για τους οικονομολόγους που αναλύουν την κατάσταση παγκοσμίου φήμης το γεγονός πως μπόρεσε να έχει τόσο καλές οικονομικές επιδόσεις η Γερμανία, πολύ καλύτερες από άλλα κράτη και γιατί ε, μπορεί να, και αυτό οφείλεται στο ότι μπόρεσε να τηρήσει δημοσιονομικούς κανόνες και προδιαγραφές, οι οποίες να δεν είναι και λάθος, ε, και να εξασφαλίσει μια, ε, ένα καλό ε, οικονομικό επίπεδο. Εγώ είμαι χρόνια τώρα πια υπουργός οικονομικών, είχα ένα ποσοστό 80% στο ε, δημόσιο χρέο τον ανέλαβα, τώρα το έχουμε κατεβάσει κάτω από το 58%, δηλαδή χαμηλότερο από το 60% που είναι το όριο του Συμφώνου Σταθερότητας και νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή επιλογή. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε την εμπιστοσύνη ότι τηρούνται οι κανόνες, μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Βέβαια, έχουμε και τη μεγαλύτερη ζήτηση ταυτόχρονα στη Γερμανία. Τη μεγαλύτερη από δεκαετίες τώρα. Μια μακροπρόθεσμα λοιπόν στεναρή, σταθερή δημοσιονομική πολιτική σημαίνει ότι ο επενδυτής και ο καταναλωτής δείχνουν εμπιστοσύνη στην οικονομία και αυτό είναι το ζητούμενο. Το καλύτερο μέσο, μέσο πρόθεσμα, είναι η αξιοπιστία. Βεβαίως και έχουν διαφορετικές οικονομικές συνθήκες στα διάφορα κράτη. Άλλα κράτη μπορεί τώρα όπως το δικό μου να έχουν λιγότερα προβλήματα από κάποια άλλα και σε αυτά τα κάποια άλλα θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη κατανόηση βεβαίως στη διαχείριση των προβλημάτων. Τους ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη σημασία. Πόσο σημαντικές είναι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Για πολλούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντικές και μάλιστα είναι κάτι το οποίο δεν συνδέεται με κάποιες εθνικές καταστάσεις και μεταρρυθμίσεις αλλά μπορούμε να πούμε με γενικό τρόπο ότι θα πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται ακόμα και οι μισθοί και σε επίπεδο επιχείρησης γιατί αυτό θα αυξήσει την προσωπική εμπλοκή του εργαζομένου και την παραγωγικότητα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσης ή αμέσως μετά από κρίση θα πρέπει να ρυθμίσουμε εκ νέου τις οικονομίες μας σε ένα εντελώς διαφορετικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε τα μέσα τα οποία να στηρίζουν τους εργαζομένους και όχι τις θέσεις εργασίας. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται σωστά οι δημοσιονομικοί πόροι. Και υπάρχει ακριβώς εδώ και η σχέση ανάμεσα ε, στις μεταρρυθμίσεις ε, και τη σύνθεση του προϋπολογισμού. Και θα πρέπει ακριβώς ε, οι δημοσιονομικές ρυθμίσεις να είναι φιλικές για την ανάπτυξη και τα μέσα, τα περιορισμένα, τα δημοσιονομικά που υπάρχουν να συνδέονται άμεσα και κυρίως με τις μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι τα βασικά θύματα της κρίσης είναι οι νέοι. Η ανεργία των νέων είναι η βασική πρόκληση. Πραγματικά κινδυνεύουμε να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά εδώ. Και γι' αυτό κάθε προσπάθεια για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης πρέπει να έχει στο νου της τους νέους. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας αυτές είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι μοναδικές, δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό πρέπει να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και στην αγορά των προϊόντων και στις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι ικανές να προσλαμβάνουν όταν υπάρχουν ευνοϊκές επενδυτικές συνθήκες. Και στο τέλος τίθεται και το θέμα της παιδείας. Νομίζω ότι βασικός οδηγός της ανάπτυξης στις προχωρημένες οικονομίες είναι οι ικανότητες και η γνώση. Ε, και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και στη δική μου κυρίως χώρα για να βελτιώσουμε το σύστημα. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν στον τομέα της παιδείας είναι συμπληρωματικές σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βλούκε για τους συντηρητικούς. Καλημέρα σας κύριε Υπουργή. Κύριε Παντοάν, η ερώτηση προς εσάς είναι πολύ σύντομη. Ο κύριος Σόιμπλα μας παρουσίασε τη Γερμανία ως υπόδειγμα στην Ευρωζώνη. Ερωτώ, λοιπόν, εσάς κύριε Παντουάν, μπορεί να ακολουθήσει και πρέπει να ακολουθήσει η Ιταλία το γερμανικό παράδειγμα. Κύριε Σόιμπλε, είπατε πολύ σωστά ότι ο απολογισμός ε, του, της κατεύθυνσης ε, της καθοδήγησης οικονομίας και το παραδέχθηκε ο συνάδελφος ομολογός σας, ε, δεν επέτυχε. Τι ήταν αυτά λοιπόν τα οποία παραγνωρίστηκαν ως στοιχεία. Ο στόχος του 3% για το έλλειμμα ε, παραβιάστηκε κατά, 90, το τελευταίο χρόνο 90 φορές. Ανταυτού όμως λέτε κοιτάμε τα διαρθρωτικά ελλείμματα και αρχίζουμε να δείχνουμε περισσότερη ευελιξία. Ωστόσο, η συμφωνία για τη μείωση των ισοτικών ελλημάτων αφορά 111 υποθέσεις παραβίασης των κανόνων που έχω καταμετρήσει εγώ, χωρίς συνέπειες, χωρίς κυρώσεις. Και άρα το ανώτατο όριο του χρέους, του 60% που έχουμε συμφωνήσει, έχει μετατραπεί σε κατώτατο όριο χρέους. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης είναι και στο 80% αλλά ακόμα και σε διπλάσια ποσοστά χρέους. Άρα και η Ιταλία τώρα και η Γαλλία βρίσκονται σε κατάσταση παραβίασης των όρων του ε, Συμφώνου Σταθερότητας, χωρίς κυρώσεις. Τώρα όμως μας λέτε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τη σταθερότητα του ε, Συμφώνου για να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να αφήσουμε τώρα κύριε Σόιμπλε οικονομικά, την, την οικονομική επιχειρηματολογία και να μιλήσουμε για μια νομική επιχειρηματολογία. Έχει διαπιστωθεί και έχει δηλωθεί και από τον το δικαστήριο της Γερμανίας ότι μπορεί να ε, αποχωρήσει από την Ευρωζώνη η Γερμανία από την ε, Ευρωζώνη στο βαθμό που αυτή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα και την οικονομία της Γερμανίας. Μπορείτε λοιπόν να συμφωνήσετε αν υπάρχει λόγος να υλοποιηθεί αυτή η προοπτική. Απάντησε κύριε κύριος σας ευχαριστώ αν θα πρέπει η Ιταλία να ακολουθήσει το άλλο παράδειγμα. Κοιτάξτε, αν πάτε πίσω 15 χρόνια, περίπου στην αρχή της Ευρωζώνης, εκείνη την περίοδο εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία είχε μπει στην Ευρωζώνη ε, σε επίπεδο ανταγωνιστικότητα σε κακή κατάσταση είχε πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα εκπέμψη χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Από τότε όμως έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο και αυτό επέτρεψε στη Γερμανία να έχει πολύ καλές επιδόσεις σε επίπεδο ανάπτυξης και σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ακόμα και στις αρχές της περίοδου ύφεση. Αυτό δείχνει ότι αν οι δομές και οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά είναι σε καλή κατάσταση τότε ε, η οικονομία θα αντέξει πολύ καλύτερα επιθέσεις όπως αυτές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσω της οικονομικής κρίσης. Ε, προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε από το παράδειγμα αυτό. Δεν είμαι απελπισμένος σε σχέση με τη δική μου χώρα. Ίσως σε λίγο χρόνια θα δούμε ότι ο κύκλος ε, της Ιταλικής ανταγωνιστικότητας θα ακολουθήσει τη σωστή πορεία. Αν τώρα κατάλαβα καλά αυτό το οποίο είπατε, Αναφερθήκατε και στις παραβιάσεις ε, των κανόνων σε σχέση με το χρέος. Ε, δεν ξέρω, ίσως σας παρανόησα, αλλά να σας θυμίσω ότι η Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι στο θέμα, στον τομέα της πρόληψης και όχι τόσο ε, στον τομέα της επιβολής κυρώσεων. Παρά το πάρα πολύ υψηλό χρέος, το οποίο είναι σημαντικό πρόβλημα και το οποίο προσπαθούμε εμείς ε, με κάθε τρόπο να κατευθύνουμε σε πτωτικές τάσεις και μέσω των, της εξυγίανσης των δημοσιονομικών πολιτικών και μέσω των μέτρων για την ανάπτυξη και κυρίως μέσω των διαφορετικών παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν στην βιωσιμότητα του χρέους αυτό. Ε, κοιτάξτε, όταν λέτε η Ιταλία παραβιάζει τους κανόνες, παρακαλώ να είστε προσεκτικός. Δείτε τους αριθμούς πρώτα. Θέλω να σας πω Καταρχά, ότι ε, μακριά από μένα η αδίποτε σκέψη να υποδείξω τη Γερμανία ω υποδειγματική περίπτωση, ω παράδειγμα προ μίμηση. Δεν είπα τίποτα τέτοιο εγώ. Μην, μην το κάνουμε αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Το πώς ρωτάτε εσείς ερωτήσεις σας είναι δική σας υπόθεση, αλλά δική μου υπόθεση είναι και το αν και το πώ θα απαντήσω εγώ στι ερωτήσει σας. Γι' αυτό μην μου υποδεικνύετε να, απαντήσω, να μην απαντήσω μόνο με ναι, να απαντήσω μόνο με ναι ή όχι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη Γερμανίας έχει μεγάλη, με μεγάλη προσοχή τηρήσει του όρου του συντάγματος, της νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένας ε, καμία περίπτωση να διαπιστωθεί παραβίαση αυτών των όρων από την τραγική ιστορία που έχουμε. Έχουμε διδαχθεί ότι πρέπει και βέβαια από δημοκρατικά νομοποιημένα όργανα να δεχόμαστε, όπως είναι το Σταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, να δεχόμαστε τον έλεγχο της στήρησης των κανόνων του συντάγματο τη νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουμε διδαχθεί από την ιστορία μα και η δική μου γενιά τουλάχιστον έχει αποκομίσει το δίδαγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το δόγμα αυτό και ελπίζω και οι επόμενες γενιές να το αποκομίσουν. Δεύτερη ερώτηση. Η Γερμανία εποφελείται όπως και κάθε άλλο κράτος από την παρουσία της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μην θεωρήσει κανείς ότι είναι ε, μία, ένα άθροισμα με μηδενικό αποτέλεσμα η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Κάθε κράτος το κάθε ένα με τον τρόπο του εποφελείται από την παρουσία του, άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο βεβαίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να κάτσω τώρα να μιλήσω για τα αδύναμα σημεία της οικονομίας της Γερμανίας, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα στα οποία έχουμε προχωρήσει και υπάρχουν και άλλα στα οποία μπορούμε να διδαχθούμε από τους εταίρους μας, τα άλλα κράτη-μέλη. Όπως μπορούμε και εμείς να δώσουμε παράδειγμα σε κάποιους άλλους, ε, όπως παραδείγματι στο σύστημα της διαδική. Εκπαίδευση που έχουμε, θεωρητική και πρακτική, δηλαδή, το οποίο φαίνεται να δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Για την ε, δημιουργία ε, ενός συστήματος σχεδιασμού για τις ε, θέσεις ε, στις αεροπορικές μεταφορές, σε παραδείγμα, μπορούμε να δεχθούμε από άλλες ε, χώρες, από άλλους εταίρους, αλλά πάλι θα καταλήξω στο συμπερασμό, στο, στη δήλωση ότι είναι κοινή ευθύνη όλων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάθε γενιά, ξέρετε η δική μου γενιά αυτό χαρακτηρίζεται ως μεταπολεμική γενιά. Εν πάση περιπτώσει είναι η γενιά η οποία προκύπτει μετά ή πάνω στα συντρίμια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και της τραγωδίας του Auschwitz η οποία εορτά, της οποίας ε, η τελική ημέρα εορτάζεται σήμερα και θέλω να σημειώσω ότι σε ένδειξη σεβασμού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθα σήμερα εδώ να σας μιλήσω αντί να είμαι στο Bundestag για, τους, ε, για την επέτειο του ε, Auschwitz. Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε γενιά μπορεί και πρέπει να διδάσκεται από την ιστορία της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εκ μέρους των φίλων ελευθέρων, κύριος Φόιερ είναι ο σκέφτης ηγετής. Α, συγγνώμη, Σοφία Ιντφελτ. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη γιατί αποσιάζει ο συνάδελφος. Είχε ενηλυμένες υποχρεώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς ε, για τις εισαγωγικές τους ε, παρατηρήσεις. Κύριε Πάντοβαν, μιλήσατε για αμοιβαία, αμοιβαίο σεβασμό. Φιντούτσα ρετσίπροκα είπατε. Αμοιβαίο σεβασμό, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό είναι από τα θεμελιώδη σημεία, τα σημεία κλειδιά. Γιατί πολλή λόγος γίνεται για αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό. Παρόλο που δεν το λέμε τόσο αναλυτικά. Μιλούμε για αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και το είναι η βάση για την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είναι όμως σημαντικό να εφαρμόζουμε ισότιμα τους κανόνες ε, ε, όλοι, να μην υπάρχουν διπλά, μέσα και σταθ, διπλά μέτρα και σταθμά, γιατί αν έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά καταργείται η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Επίσης θα πρέπει να μιλάμε με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον και να αποφύγουμε τις καρικατούρες γιατί και η ψυχολογική διάσταση παίζει μεγάλο ρόλο στην ε, εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και να κάνουμε ό,τι λέμε. Γιατί πολλές φορές στο Συμβούλιο ακούμε δηλώσεις για τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη σημασία της εσωτερικής αγοράς, τη σπουδαιότητα των επενδύσεων. Διαπιστώνω όμως ότι το ίδιο το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη, δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Πολλά λόγια ακούμε για την εσωτερική αγορά, αλλά το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες βρίσκεται ακόμη σε αποτελμάτωση. Μιλούμε για επενδύσεις, αλλά μέχρι στιγμής τα κράτη-μέλη απέτυχαν να, να πλήρω πλήρως το επενδυτικό πακέτο και άλλες δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί δεν έχουν εφαρμοστεί. Πώς λοιπόν θα περάσουμε από τη φάση των λόγων στη φάση των έργων, και τι θα κάνετε όχι μόνο για να εξασφαλίσετε δημοσιονομική πειθαρχία αλλά και την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς και την υλοποίηση του επενδυτικού πακέτου που χρειαζόμαστε καταπηγόντως. Σε ποιο πακέτο αναφερθήκατε, ποιο πακέτο λέτε ότι δεν εφαρμόστηκε. Α, των τηλεπικοινωνιών. Αναφέρθηκα στο πακέτο των τηλεπικοινωνιών και την ε, ε, έλλειψη ακόμη δέσμευση υπέρ του επενδυτικού πακέτου εκ μέρου των κρατών μελών. Δεν είναι τόσο ερώτηση. Είναι μια δήλωση περισσότερο αυτό που κάνατε και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να απαντήσω. Αλλά σταθώ σε ένα σημείο το οποίο ε, έχει σημασία. Πρόκειται για το επενδυτικό πρόγραμμα. Έχω την αίσθηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και όχι μόνο γιατί έχει παρουσιάσει απλά αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα ο πρόεδρος Γιούνκερ το οποίο αρχίζει και αποκτά λεπτομέρειες σε σχέση με τους πόρους και την αρχιτεκτονική του. Αλλά και εδώ ε, ο ομιλός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης κράτους μέλους, ε, αλλά ε, αυτή η πρόταση αλλάζει και τις προοπτικές με τον τρόπο, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας η επένδυση, οι επενδύσεις είναι το βασικό χαρακτηριστικό ε, επηρεασμού της οικονομικής ανάπτυξης. Ξέρετε ότι έχουν μειωθεί οι επενδύσεις όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο μετά από την αρχή της κρίσης και πρέπει να αναζωογονήσουμε τις επενδύσεις όχι μόνο για να υπάρξει ανάκαμψη βραχυπρόθεσμη της ζήτησης αλλά να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τις οικονομίες μας την ανάπτυξη, ε, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κτλ. Λοιπόν, τι έχει αλλάξει. Το θέμα δεν είναι να συζητήσουμε απλά την αρχιτεκτονική ε, του συγκεκριμένου αυτού του στρατηγικού επενδυτικού ταμείου, αλλά για να υπάρξει ανάκαμψη της επένδυσης απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, απαιτούνται πόροι και φυσικά και πόροι από πλευράς του δημοσίου τομέα αυτό είναι πιο σημαντικό, ιδιαίτερα για τη μόχλευσή τους που θα οδηγήσει και σε επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Και δεύτερον, οι πόροι αυτοί θα πρέπει να καλύψουν ανάγκες οι οποίες είναι ε, επενδυτικά βιώσιμες. Και πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και την προγραμματική δυνατότητα, αν θέλετε, και των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά ε, και των ε, ιδιωτών που επιζητούν χρηματοδοτήσεις. Οι κυβερνήσεις λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν και υποβάλλουν αιτήσει για χρηματοδότηση προγραμμάτων. Και γι' αυτό ακριβώς η Task Force που δημιουργήθηκε το προηγούμενο εξάμεινο ήδη έχει ε, δώσει κάποιες, κάποιους καρπούς οι οποίοι πρέπει να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας περαιτέρω. Πάντως το θέμα με τους δημόσιους πόρους δεν είναι αν είναι πολύ λίγοι, το θέμα είναι κυρίως να δούμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν και θα βελτιωθούμε έτσι την αποδοτικότητα των επενδύσεων και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο. Κύριε Νιτφέλτ, νομίζω ότι με τις επενδύσεις το πρόβλημα είναι όχι μόνο να υπάρχουν τα διαθέσιμα μέσα αλλά και να υλοποιούνται. και αυτό τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και έδωσα ένα παράδειγμα από τη δική μου πατρίδα ότι χρειαζόμαστε δηλαδή καλύτερη και πιο αποτελεσματική υλοποίηση για το πακέτο των τηλεπικοινωνιών θεωρώ γιατί συνομιλήσαμε ακόμη την Κυριακή το βράδυ με τον Επίτροπο Ετιγκέρη ότι, είναι πολύ, κοντά η υποβολή από πλευρά του των προτάσεων. Και έτσι τίθεται το ζήτημα πλέον της ευρωπαϊκής Ρύθμιση με βάση το Ευρωπαϊκό Πρωτογενέ Δίκαιο. Και βεβαίω τώρα πρέπει να προχωρήσουμε προ μια απορρίθμιση. Αυτό χρειαζόμαστε. Και έτσι με την ε, ε, Προεδρία του Πιέρ Κάρλο Πάντοαν στι ε, αρχέ Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο των Υπουργών των Οικονομικών σε ένα άτυπο συνέδριο στο Μιλάνο, άτυπη συνάντηση στο Μιλάνο, είπαμε ότι θέλουμε για του νέου να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση και επενδύσει, αλλά όχι σε όρου τι χρήμα ρίχνω, αλλά σε όρους βιώσιμης επένδυσης. Και γι' αυτό μιλήσαμε για μια τράπεζα επενδύσεων που μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαληθεύει ότι υλοποιούνται οι επενδύσεις και όχι ότι ρίχνουμε μόνο νούμερα πάνω στο τραπέζι, χωρίς αποτέλεσμα. Για να μπορούμε μέσα σε ένα χρόνο να λέμε ότι να υπάρχουν αποτέλεσματα. Ε, εκεί πρέπει τα χρήματα πράγματι να αξιοποιούνται σωστά. Οι πόροι να χρησιμοποιούνται για να ενισχύουν τις δομές στα κράτη-μέλη. Αυτό γίνεται και στην Ευρώπη, πρέπει να γίνεται και σε εθνικό επίπεδο. Και εμείς και στη Γερμανία κάνουμε ό,τι μπορούμε με το περιθώριο που έχουμε για να προσελκύσουμε πρόσθετες επενδύσεις. Μη συμφωνούμε σε αυτό, στον κυβερνητικό συνασπισμό, και άλλωστε έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να προσελκύσουμε σωστές επενδύσεις και για τη Γερμανία. Ευχαριστώ. Αρχίζει και μας πιέζει ο χρόνος. Τώρα θα ομοδοποιούμε τις ερωτήσεις. Ο Φάμπι Ντεμάζη από την ΚΟΕ. Κύριε Σόιμπλε, καλημέρα. Σας μιλήσατε για την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ε, θεωρώ ότι η πολιτική ηγεσία στις κυβερνήσεις της ε, Ευρώπης θα όφιλε να διαρωτηθεί περισσότερο για την εμπιστοσύνη ότι έχει των χρηματοπιστωτικών αλλά της μεγάλης πλειονοψηφίας των λαών της Ευρώπης. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό να το λησμονούμε και θα πρέπει να κοιτάμε τα γεγονότα. Η Ευρώπη είχε με στοιχεία του ΩΣΑ ένα από τα πιο σκληρά πακέτα προσαρμογής για κράτος βιομηχανικό μετά στη μεταπολεμική ε, περίοδο. Το χρέος της αυξήθηκε από το 130% στο 170%. Η ανάπτυξη έχει καταρρεύσει. Η ανεργία κυρίως των νέων είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Και σε αυτό μπορεί να έχετε τη της Ελλάδας. Και σε αυτό μπορεί να έχετε διαφορετική εκτίμηση ίσως, αλλά έχουμε στοιχεία από την κεντρική τράπεζα, κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα, η οποία λέει ότι μπορεί και για το σύστημα της ε, κατεπίγουσας ε, ε, ενίσχυσης για τη ρευστότητα να δώσει κάποια λύση ε, με ε, περιορισμένες αγορές ομολόγων. Θεωρείται λοιπόν ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις θέσεις, με τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και σε περίοδο κρίση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ε, δέχεται ε, χρεόγραφα από ιδιωτικού φορεί. Και δεύτερον, μιλήσατε για διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Χρειάζεται όντω η Ελλάδα διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Αλλά γιατί η γερμανική κυβέρνηση επιμένει να μην ε, πιέζει για περισσότερη ε, φορολόγηση ε, των επιπέδων περιουσιών, όπως πιστεύω ότι θα έπρεπε να συμβαίνει. Ο κύριος Φίγκολτ έχει το λόγο. Το ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης το συζητούμε εδώ. Έχουμε τους υπουργούς των οικονομικών της ε, Ιταλίας και της Γερμανίας που νομίζω ότι συμβολικά εκπροσωπούν και τον τύπο των προβλημάτων που συναντούμε στην Ευρώπη. Εσείς στην Ιταλία έχετε ε, διέλθει μια πολύ σκληρή περίοδο κρίσης με πολύ σημαντική πτώση της ζήτησης ενώ η Γερμανία με χαμηλά επιτόκια μπόρεσε να έχει ε, στο χώρο των δημοσιονομικών της σημαντικό περιθώριο ελιγμών να περιορίσει το χρέος της, να προχωρήσει με το σύστημα του εξάπτυχου σε σημαντική μείωση του χρέους και έτσι τίθεται το ερώτημα. Τώρα η Ιταλία παραμένει ε, μια χώρα με σημαντικά προβλήματα ζήτησης. Μπορεί η Γερμανία να στηρίξει την Ιταλία σε αυτό. Και επίσης κύριε Σόιμπλε, πολλές από τις ε, δεσμεύσεις της Γερμανίας για το δημοσιονομικό συντονισμό δεν έχουν τηρηθεί. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό ο δημοσιονομικός συντονισμός λοιπόν κύριε Σόιμπλε. Και εσείς κύριε Παντοάν ε, πώς κρίνετε τη δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας. Θεωρείτε, ότι θα πρέπει να έχει μια πιο ανοιχτή πολιτική με πιο πολλές επενδύσεις που να αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών ώστε να μην ε, ε, διαιωνίζεται μια κρίση και εσείς κύριε Σόιμπλε γιατί θεωρείτε ότι πρέπει με τα σχέδιά σας να επιβάλλετε υπερβολική τήρηση των κανόνων και όχι μόνο στη Γερμανία και γιατί να μην δώσουμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο και στους εταίρους μας της Ευρώπης ώστε να δούμε στο μέλλον ένα εσωσκελισμό, μια εξισορρόπηση των ε, δημοσιονομικών αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ κύριος Μαρκοβάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημερίζω λοιπόν τους δύο υπουργούς. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο ε, κυρίως προς τον Γερμανό Υπουργό ε, ξέρετε ότι πολλά πράγματα καθορίζονται από την Τρόικα, την οποία ποτέ κανένας δεν ψήφισε βέβαια μέχρι τώρα. Θα ήθελα να μάθω αν στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες τάσεις για αλλαγές που θα οδηγήσουν σε μια αντιμετώπιση των προβλημάτων με πιο ειρηνικό τρόπο ή θα επιμείνετε με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο ε, στα δημοσιονομικά μέτρα και στη δημοσιονομική εξυγένση. Ε, με τις αιμονές ε, σας αυτές έχετε καταστρέψει το ευρώ, έχετε καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε δεκάδες πολύ γνωστών οικονομολόγων σε όλο τον κόσμο. Οι διαδικασίες για το ευρώ θα έπρεπε να είναι διαφορετικές. Όλα αυτά όμως απέτυχαν και αποτύχατε. Γιατί δεν βάζετε στο κέντρο ε, της ε, προσπάθειά σας την προάσπιση των συμφερόντων των πιστοτικών οργανισμών και όχι την αλληλεγγύη των λαών, όχι την αλληλεγγύη με τους λαούς του Νότου αλλά κυρίως την αλληλεγγύη με τις πολιεθνικές του Λουξεμβούργου επί δεκαετίες και μετά από ε, αυτές όλες οι δηλώσεις οι απειλητικές των αρχηγών κυβερνήσεων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς την Ελλάδα δεν έπρεπε να είχαν την Ελλάδα παραλήπτη αλλά το Λουξεμβούργο. Λοιπόν με τη λογική σας και τις αιμονές σας η Ευρώπη ε, έχει αρχίσει να ε, φτωχαίνει. Εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε το πρόγραμμα Quantitative Easing το οποίο δεν έχει της ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο δεν έχει ε, παρά αποδείξει ε, ότι τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα ε, σοβαρά. Η Γερμανία βέβαια την χάνει να βρίσκεται σε μια κατάσταση εποφελούμενη από τη σταθερότητα του ευρώ και η Γερμανία είναι ίσως και η μόνη που ωφελείται από αυτό. Who wants to start? Ο λόγος καλεσμένος μας. Ποιος θα αρχίσει? Απαντήστε συνολικά και στις τρεις ερωτήσεις. Κύριο Σουέμπλε. Δεν θα είναι εύκολο κύριε Πρόεδρε. Να, ήταν πολλές οι παρατηρήσεις και λίγες οι ερωτήσεις. Κάτι το οποίο είναι και συνηθισμένο στην πολιτική η έκθεση διαφορετικών προοπτικών και τοποθετήσεων. Αλλά μην περιμένετε να απαντήσω με τους δικούς σας όρους. Θα κάνω όμως την παρατήρηση, κύριε συνάδελφε, πρώτον ότι δεν σχολιάζω ως υπουργό των Οικονομικών αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία φέρει την ευθύνη για την νομισματική πολιτική, η οποία είναι ανεξάρτητη και για πολύ σοβαρούς λόγους, και ως εκ τούτου οφείλουμε να δεχόμαστε, να αποδεχόμαστε τις αποφάσεις της. Δεν αποφασίζει ένα υπουργό οικονομικών, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα για την νομισματική πολιτική. Ο Μάριο Ντράγκη το λέει και το επαναλαμβάνει διαρκώ ότι χρειάζεται όμω και μια υγιή οικονομική διαχείριση. Έχουμε να κάνουμε με ένα τρίπτυχο που είναι τα κράτη, με τι εκλεγμένε κυβερνήσει, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και βεβαίω με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ελλάδα, αυτό που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ως προϋπόθεση είναι απόλυτο σύμφωνο με, με τη βασική της γραμμή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε γι' αυτό και, διάβασα πολύ προσεκτικά, καμία σχέση δεν έχει με τις παρατηρήσεις, με τις προτάσεις ε, του εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό που είπατε δεν είναι αληθές δηλαδή. Επίσης για την Ελλάδα έχω να πω ότι η Ελλάδα εψήφισε, ήταν σαφέστατο το αποτέλεσμα της Κυριακής, σχηματίστηκε ένας ενδιαφέρον συνασπισμός, δίπλα-δίπλα κάθονται, πολύ ωραία, αξιόλογα, αξιο... άξιο τους δώσουμε προσοχή δεν λύνονται όμως έτσι τα προβλήματα της Ελλάδας. Ο ελληνικός λαός υποφέρει περισσότερο από ό,τι άλλα κράτη. Τα κράτη τα οποία βρέθηκαν, ε, ε, ήταν μέχρι το 90 στην ε, ηγεμονική, στον ηγεμονικό χώρο του σοσιαλισμού, η κατάσταση μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, αλλά η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην κατάσταση αυτή γιατί φταίνε οι Βρυξέλλες ή η Ευρώπη κάποιος άλλος, αλλά γιατί και οι πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας έκαναν λάθος επιλογές για πολλά χρόνια. Και έτσι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Το να συζητούμε ότι χρειάζεται να ληφθεί μια διαφορετική απόφαση είναι χάσιμο χρόνου. Εγώ ως Υπουργό των Οικονομικών της Γερμανίας μαζί με τους άλλους υπουργού Οικονομικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια για τη στήριξη της Ελλάδας, η οποία Ελλάδα αξιοποίησε περιορισμένα μόνο αυτή την προσφορά βοήθειας, αλλά οφείλουμε να το σεβαστούμε. Για τα γερμανικά, γερμανογερμανικά θέματα, αγαπητέ φίλε και συναδελφέ, δεν χρειάζεται να συζητούμε γιατί δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι έχουμε λιγότερο χρέος, υψηλότερη ανάπτυξη από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα κράτη τα οποία έχουν περάσει από προγράμματα προσαρμογής, τα πέντε αυτά του ΩΣΑ που καταγράφει στην έκθεσή του για τα πέντε κράτη τα οποία είχαν τις καλύτερες επιδόσεις με τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα πρώτα απ' όλα, μη ότι δεν ήταν σε καλό δρόμο το πρόγραμμα, γιατί και η Ελλάδα μπόρεσε να έχει, να για πρώτη φορά πρωτογενές πλεόνασμα και τώρα έχει μπροστά, ακόμα, μπροστά του ακόμα ο ελληνικός λαός ένα σκληρό δρόμο αλλά έχει μπει στο σωστό δρόμο και το λέω αυτό εξ αρχής και ως υπουργό των οικονομικών της Γερμανίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στη μόνη ερώτηση που αν δεν κάνω λάθος απευθυνόταν σε μένα. Ε, με ρωτήσατε πιστεύω ότι οι περισσότερες επενδύσεις θα κάνουν καλό και στην Γερμανία. Δεν είναι κάτι καινούριο και οι γερμανικές αρχές και φαντάζομαι θα συμφωνήσει και ο Βόλφκανγκ. Το θέμα δεν είναι αν χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, αλλά από πού θα προέλθουν αυτές και πώς θα ενεργοποιηθούν. Συμφωνώ με αυτό που λένε όσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επαριλημμένος, ότι πολλές χώρες έχουν ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το ίδιο και η Γερμανία και κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθούν οι επενδύσεις από περαιτέρω απελευθέρωση κάποιων κλάδων που θα τονώσουν τις ε, ιδιωτικέ επενδύσει. Ό,τι αφορά τι ε, δημόσιε επενδύσει, η γερμανική κυβέρνηση ήδη έχει ξεκινήσει ένα σχετικό πρόγραμμα, οπότε ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα αποβεί προ όφελο και τη Γερμανία και ολόκληρη τη Ευρωζώνη εξαιτία τη αλληλεπίδραση ε, και θα διορθώσει και κάποιε ανισορροπίε. Ευχαριστώ. Μα έμεινε ένα λεπτό ακόμη για την εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς ε, για την ανταλλαγή απόψεων που κάναμε. Πολλά υπόθηκαν και για τη φύση των διαστρωτικών μεταρρυθμίσεων και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν στον κύκλο της οικονομικής διακυβέρνησης. Και θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει συζήτηση για το τι θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο και τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σεβασμό των κανόνων ή με την προοπτική κάποιας αλλαγής τους. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γενική κατάσταση της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την ικανότητά της να αντιμετωπίσει σύσσωμη τις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας. Κύριε Σόιμπλε, είπατε ότι θα πρέπει να βρούμε συμφωνίες για μεταφορές και αντισταθμίσεις. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και σίγουρα αυτό το δρόμο, αυτή την πρόταση θα πρέπει να την αναπτύξουμε περαιτέρω και να δούμε και τις επιπτώσεις της ε, εντός της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας ε, και τις ε, παρατηρήσεις σας. Φαντάζομαι θα υπάρξει συνέχεια και διαλληλογραφίες για να μπορέσουμε στο δεύτερο τρίμηνο να αποκρισταλώσουμε τη θέση μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την αξιολόγηση της ευελιξίας και για το περιθώριο ελιγμών που αφήνουν οι αξιολογήσεις ε, του εξάπτυχου και του δίστυχου πακέτου και την αξιολόγηση που θα κάνουμε της έκθεσης των τεσσάρων προέδρων. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους μας. Πολύ ενδιαφέρουσα και καρποφόρα η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Να σας υπενθυμίσω τα επόμενα βήματα της έκτης Μπερές. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης 23 και 24 Φεβρουαρίου, προθεσμία για τις τροπολογίες 3 Μαρτίου, εξέταση των τροπολογιών 23 και 24 Μαρτίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 14 ε, Απριλίου και στη δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου θα εξεταστεί η έκθεση αυτή. Αυτά λίγε η συνεδρίαση. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσει η συνεδρίαση σε 5 λεπτά με το σημείο 8 της ημερησίας διατάξεως και προεδρία του κυρίου Φέρπερ. So, dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ, όσοι έχουν άλλα αναπόδραστα καθήκοντα, ας αποχωρήσουν για να τα εκτελέσουν και να συνεχίσουμε στη δουλειά μας. Ναι. ναι, σοβαρή δουλειά κάνουμε εμείς εδώ. Δεν ξέρω οι άλλοι τι μερίσια διάταξη έχουν, εμείς πάντως έχουμε σοβαρή δουλειά. Δεν μπορώ να αξιολογήσω τη δουλειά των άλλων. Αυτά λοιπόν. Πρώτον, ανακοίνωση για το απόγευμα. Υπενθυμίζω ότι από τις 3 έως τις 3.30 το απόγευμα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση έκον και λίμπε στην ίδια για να αξιολογήσουμε την έκβαση των διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου για την ε, νομοποίηση παρανόμων εσόδων Παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι θα υπάρξει διαφορετική ρύθμιση ως προς τις θέσεις που κάθεστε κανονικά, μια και θα είναι μεικτή η συνεδρίαση, κοινή συνεδρίαση. Μην αφήσετε κάρτες ψηφοφορίας, μην αφήσετε κινητά. Θα είναι διαφορετική η σύνθεση της ε, αίθουσας την ώρα που θα γυρίσετε το απόγευμα. Και τώρα έχουμε τον έλεγχο των ακροπεξουσιοδότων συμπράξεων και των εκτελεστικών μέτρων, σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη. και εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε τα μέτρα που έχουν προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε τις αρχές, τις εξουσίες που έχουμε για ε, επισκόπηση αυτής της ε, κατάστασης. Η Τραπεζική Αρχή Εποπτείας έχει ορίσει μη δεσμευτικά επίπεδα κάτω από τις κατεξουσιοδότηση πράξει και εκτελεστικά μέτρα. Ωστόσο, εμεί ασκούμε ω Επιτροπή των Οικονομικών ε, τι αρμοδιότητέ μα και στι 11 Νοεμβρίου του 2014 ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών ε, με ένα έγγραφο για τα συστήματα εγγύσεων υπό το άρθρο 3 της σχετικής οδηγίας μια πρόταση που μπορούμε να τροποποιήσουμε μέσα στον Φεβρουάριο. Ο κύριος Τζασκαρόν από την EBA είναι εδώ, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Τον καλωσορίζω, τον παρακαλώ να μας ενημερώσει για το θέμα αυτό και μετά την εισαγωγή θα συζητήσουν πρώτα οι συνάδελφοι συντονιστές και μετά η λοιποί με τη διαδικασία ΚΑΡΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Κανόνα έχει το λόγο λοιπόν. Thank you very much. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για την αλλαγή απόψεων στα πλαίσια του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις κατεξιδότητες πράξεις και για, για τις κατευθυντήρες γραμμές. Τα κράτη-μέλη έχουν λίγους μήνες ακόμη πριν τη λήξη της προθεσμίας ενσωμάτωσης της νέας αυτής οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ε, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία με συμβολές, με δεσμεύσεις πληρωμών και με τα stress test και κάποιες συμφωνίες συνεργασίες. Είναι σημαντικές λοιπόν, ε, σημαντική συνεισφορά μας. Η πρόκληση ήταν να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ ενός ε, τεχνικός υγιούς πλαισίου και αφετέρου της δέουσας ε, σύγκλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των τραπεζικών μοντέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ε, τεχνική αρτιότητα, νομίζω ότι έχουμε ένα πλαίσιο που έχει σωστά χρονοδιαγράμματα το 2024 και σωστό επίπεδο στόχων και δίνουμε κίνητρα για σωστή συμπεριφορά απέναντι στον κίνδυνο με νέα δείκτες ε, κινδύνου που καλύπτουν τις βασικές θεραπευτικές δραστηριότητες, ε, ποιότητα τίτλων και περιουσιακών στοιχείων, ποιοτικό management και το καθεξής. Οπότε θα πρέπει, δίνονται κάποια στοιχεία για το πώς θα μπορέσει να επέμβει η DGS σε περίπτωση χρεοκοπής και αν χρεοκοπήσει η τράπεζα, ποιο είναι το επίπεδο ζημιών που θα πρέπει να καλύψει ίσως η DGS. Θέλουμε διαφοροποίηση του κινδύνου, εξασφάλιση διαφοροποίηση του κινδύνου με ελάχιστη διαφοροποίηση μεταξύ 75% και 150% του μέσου όρου. Πάνω κάτω δηλαδή λίγο περισσότερο από ό,τι προβλέπει η καταξιδότηση πράξη για τη συμβολή στο Ταμείο Εξυγίασης. Θα θέλουμε να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ εναρμόνισης και ηθικών θεμητού ανταγωνισμού αφενό και ευελιξία αφετέρου. Και υπάρχει αρκετό περιθώριο λιγμών για τα κράτη-μέλη και, και για την DGS για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητε των μοντέλων. Επίση, αναφέρθηκε η μέθοδο του ίδιου κινδύνου και τη δυνατότητα προσδιορισμού ελάχιστη συμμετοχή ή χαμηλότερη συμμετοχή για κλάδου μικρού κινδύνου ή για τράπεζες που είναι μέλη ενός IPS. Επίσης, δυνατότητα ελεύθερης κατανομής των, του βάρους του ε, κινδύνου πάνω από 25% και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να αφαιρεθεί ένας υποχρεωτικός δείκτης ε, κινδύνου όταν δεν υπάρχει. Επίσης υπάρχει ευελιξία για τη στάθμη βαθμονόμηση των αιτιών του κινδύνου και ε, είπαμε 75 με 50% είναι το φάσμα της απόκλησης. Κατευθυντήρες γραμμές μέχρι 11 Φεβρουαρίου περιμένουμε. Ε, βέβαια τελευταία στιγμή δεν αντέει οι σχολιασμοί. Είχαμε, συναντήσεις με διαφερόμενους και διμερός, αλλά είχαμε και στις 8 Ιανουαρίου τη σχετική δημόσια ακρόση. Επί του παρόντος μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι διαφερόμενοι τάχθηκαν υπέρ του γενικού πλαισίου δεν υπάρχει φυσικά ομοφωνία, αλλά υπάρχει γενική υποστήριξη. Το θέμα είναι αν αρκεί 25% ευελιξία ή είναι υπερβολικό το ποσοστό αυτό. Δεν έχουμε καταλήξει συμπέρασμα γιατί άλλοι είναι υπέρ ποσοστού και άλλοι υπέρ Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα σοβαρό και αξιόπιστο επίπεδο συνθηκών θεμητού ανταγωνισμού και ισότιμου ανταγωνισμού. Κάτι άλλο που σας ενδιαφέρει και εσάς και το συμπεριλάβαμε στη συζήτηση είναι οι, τα κεντρικές οντότητες του IPS. Μιλούμε για ένα σύστημα θεσμικής προστασίας που μπορεί να μην αναγνωρίζεται σε επίσημο DGS, αλλά οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει πολλές μικρές τράπεζες που έχουν καταθέσεις, αλλά είναι μικρές στο μέγεθός τους και στηρίζονται σε υπηρεσίες πολύ μεγαλύτερων κεντρικών ιδρυμάτων. Οπότε εφαρμόζοντας τη μέθοδο αυτή, μας λένε μερικοί δεν μπορώ να χρεώσω μεγάλες συνεισφορές στις μεγάλες τράπεζες, γιατί οι μεγάλες ε, δεν καλύπτουν τόσο περισσότερες, τόσο μεγάλες καταθέσεις, αλλά δημιουργούν μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο. Οπότε αρχίσαμε αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη, εξετάζοντας από τη δημοσίευση τους κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να έχουμε ειδικού δείκτες για τα ιδρύματα που έχουν συστημικό χαρακτήρα εξαιτία ε, του μεγέθους τους και εδώ ε, θα έχουμε ίσως και ένα 25% του συνολικού φόρμουλας. Δεν ξέρω αν αρκεί αυτό. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε μήπως θα μπορέσουμε τέτοιες ε, περιστάσεις να τις χρεώσουμε στο δίκτυο της ελάχιστης εισφοράς. Η εδώ προσπαθούμε να καλύψουμε τις, τις καταθέσεις με aggregate ε, risk weight, με συνολικό βάρος κινδύνου. Τώρα, αν στην ελέγξη συνεισφορά έχουμε ιδιαίτερη κατάσταση, ακόμη και αν τα κεντρικά ιδρύματα έχουν ένα μικρό επίπεδο καλυμμένων ε, καταθέσεων, θα μπορούσαμε να ε, επανισορροπήσουμε τον κίνδυνό τους για το σύστημα, εξαιτίας του γεγονότος ότι το σύστημα υπάρχει, εντάσσεται στην ελάχιστη συνεισφορά. Μιλήσαμε και για τις τράπεζες τρίτων χωρών, κυρίως θηγατρικές σε τρίτες χώρες. Είναι ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με τους ενδιαφερόμενους και είμαι στη διάθεσή για περαιτέρω ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ κύριε Κανόνε. Συγγνώμη με τον εισηγητή, μετά με τους συντονιστές και στη συνέχεια η συνάδελφη. Ο Πέτρας Σιμών. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ κύριε Κανόνε για τη δεξοδική αυτή έκθεση των βασικών γραμμών, των κατευθυντήριων γραμμών ε, που έχετε υποβάλει για διαβούλευση. Ε, κοιτώντας λοιπόν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, βλέπουμε πόσες είναι οι διαφορετικών ε, τομέων που προσπαθείτε να καλύψετε και να ίσως σταθμίσετε, να εξισορροπήσετε, ώστε να εξασφαλιστεί μια καλή στάθμιση για την Ευρώπη των κινδύνων, με τη συμβολή βεβαίως των επιμέρων ε, των επιμέρους ε, οικονομικών παρεμβάσεων των ε, τραπεζών. Ένα-δύο σημεία όμως μου γεννούν μεγάλα ερωτηματικά. Τα αγγίξατε ακροθυγώς. Θα, θα τα διατυπώσω λοιπόν. Το πρώτο έχει να κάνει με το ζήτημα της ευελιξίας. Ως εισηγητής είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολλούς με εκπροσώπους συστημάτων διασφάλισης ε, καταθέσεων και με διαφορετικές απόψεις που είδα καταλήγω ότι το Κοινοβούλιο θέλει να έχει ευελιξία βέβαια μέσα σε ένα σύστημα που λειτουργεί καλά, που μπορεί να λειτουργεί καλά, το οποίο όμως δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί εκ Όταν λοιπόν λέτε ότι στην πρότασή σας έχετε 75% των δικτών παγιωμένο και 25% ευέλικτο. Το ερώτημα είναι, αρκεί αυτό το 25% της ευελιξίας. Θα μας δώσετε κάποιες περιττέρω εξηγήσεις γιατί θεωρείτε ότι μπορεί να αρκεί αυτό. Να αρκεί αυτό. Και επίσης, μια δεύτερη ερώτηση, στο πλαίσιο αυτό πάντα, εάν αυτό το 25% που χαρακτηρίζεται ευέλικτο είναι όντως ευέλικτο. Και αν κοιτάξουμε κάποια σενάρια τα οποία μας έχετε δώσει με τις κατευθυντηρίες γραμμές και την πρότασή σας με το 25% βλέπουμε ότι αυτό το 25% συνδέεται σε διάφορους όρους και προϋποθέσεις. Δεν αφήνεται δηλαδή κάποιους δείκτες ελεύθερους και ενδεχομένως σε κίνδυνο ή διακινδύνευση, αλλά ορίζεται ε, τα επίπεδα ή ε, όρια. Αυτή είναι λοιπόν κατ' επίφαση η ευελιξία κατά την υπόψη μου. Ένα στενός κορσές δηλαδή είναι αυτό που μας προτείνεται. Δεν υπάρχει περιθώριο ή και αν δεν είναι μηδενικό πάντως είναι πολύ χαμηλό το περιθώριο των ε, χειρισμών τη ευελιξία. Δεύτερον, το σύστημα διασφάλιση που αναφέρατε τα συστήματα διασφάλισης. Όπου λέτε κι εσείς ότι λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες του 64, του 65 στις σας γραμμές με τα συστήματα διασφάλισης. Πολύ σας, πολύ ωραία. ωραία. Προσθέτω αυτών των ε, συστημάτων διασφάλισης, όποιος χρειάζεται δηλαδή να προχωρήσει πέραν αυτών, μπορεί να πάρει μια έκπτωση. Έστω αλλά το τελευταίο που αναφέρατε δεν ήταν πολύ σαφές. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος μπαίνει στο σύστημα διασφάλισης και ε, αναγνωρίζεται ο ίδιος ως σύστημα διασφάλισης καταθέσεων. Τι είναι αυτός, ή μάλλον ε, σύστημα διασφάλισης των ε, πόρων, των καταθέσεων. Τι γίνεται λοιπόν αυτός. Τα κεντρικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν αυτά τα οποία στην κρίση αντιμετώπισαν τα προβλήματα και στη Γερμανία. Τα μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είχαν τόσο πρόβλημα. Τώρα λοιπόν ε, τα, με, τα μέχρι τώρα συστήματα διασφάλισης, ας κοιτάξουμε τις ε, τράπεζες Γερμανίας, έχουμε 60 πλάσια κάλυψη από την μικρή τράπεζα, αυτή που έχει λιγότερη έκθεση. Με το δικό σας λοιπόν σύστημα, με το 75-25% θα, φτάσω, θα φτάνουμε στο οκταπλάσιο. Ισοδύναμο δηλαδή κίνδυνο με αυτόν που έχουμε τώρα. Εάν αυτή η εξαίρεση που έχετε πριν το 66, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λόγια σας, πιάνει μόνο τα χρηματοπιστωτικά και είναι ιδρύματα που έχουν περιορισμένες καταθέσεις αλλά υψηλό κίνδυνο με το 25% της ευελιξίας. Μόνο 25% όμως μπορούν να έχουν. Και όχι 100% των εισφορών. Ε, αυτό δεν αρκεί. Για να ε, εξισορροπηθεί αυτός ο κίνδυνος όπως τώρα. Και σας δηλώνω ξεκάθαρα ότι έχω πολύ μεγάλη αμφισβήτηση για το αν μπορεί ε, ένας τέτοιος, ε, ένα τέτοιο σύστημα να δώσει αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, να κοιτάξετε τουλάχιστον να έχετε κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Με την έννοια ότι αυτό που μας δίδαξε η κρίση, η μέχρι τώρα κρίση, είναι ε, ότι πρέπει όχι λιγότερα ποσά διασφάλισης, αλλά περισσότερα ποσά διασφάλισης να έχουμε στη θέση μας. Πράγμα το οποίο δεν μας επιτρέπει το άρθρο 66 από ό,τι βλέπω, γιατί μόνο στο 25% μπορούμε να έχουμε ευελιξία και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας θέση. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ και αν συμφωνείτε να ακούσουμε πρώτα τους και ηγητές για να μαζέψουμε τις ερωτήσεις. Ο κύριο Μπάλτσα έχει το λόγο εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Πέτερ Ζημών για τι παρατηρήσει και ερωτήσει του. Γιατί άφησε τα ζητήματα τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εδώ. Εμένα και όλη μου την ομάδα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στη γραμμή στην οποία έχουμε συμφωνήσει την εξαιρετική ρύθμιση του άρθρου 13 παράγραφος 2 που μου φαίνεται ανεπαρκής. Πρόκειται για μια ρύθμιση εξαίρεσης λοιπόν η οποία μπορεί να επιτρέψει την ε, χρήση των μεθόδων ε, που στηρίζουν στον κίνδυνο για τα μέλη με βάση τον στόχο της ε, διασφάλισης των ε, καταθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη, και εδώ παραθέτω ρητά το άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη την ρευστότητα και το βάρος των ε, ποσών των πόρων. Εδώ όμως πρέπει να δούμε σε ποιο ε, βαθμό καλύπτονται οι καταθέσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ποιο είναι το ύψος της κάλυψης. Και ακριβώς πρέπει να δούμε τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών αυτών τα 10 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα φαίνεται να μην έχουν κανένα περιθώριο με βάση το άρθρο 13, παράγραφος 2. Αυτός είναι άλλος το στόχος του άρθρου. Το Ινστιτούτο θα πρέπει να μπορεί να συμβάλλει σημαντικά, όπως και στο παρελθόν, στην ε, σταθερότητα και στο μέλλον. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι ασφαλώς δεν μπορεί η οδηγία μας να επιδιώκει τη σταθερότητα αυτή ε, ή οι κατευθυντηρίες γραμμές της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχαίας να ε, αμφισβητούνται εν τέλει, να υπονομεύονται. Είναι απαραίτητο να μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή αρχαιης να αμφισβητουνται εν τελει να Αρχή όπου και όπως χρειάζεται και εδώ νομίζω το άρθρο 13 παράθρος 2 λέει σαφώς ότι οι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ορίζουν τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών ε, με βάση τις παραγράφους 1 και 2 προσδιορίζονται συγκεκριμονοποιούνται με βάση παραγράφους 1 και 2. Και μετά πάμε στο 13.2 με την εξαιρετική ρύθμιση. Εδώ θα ήθελα λοιπόν κάποιες σαφέστερες ε, τοποθετήσεις από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ευχαριστώ πολύ. ECR, Τσέχο. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ εδώ το σκιώδη μας ηγητή. Ο σκιώδης ηγητής μας ε, από τη CCR περιμένει τις διαβουλεύσεις για τις κατευθυντήρες γραμμές. Είμαστε υπέρ των συνεισφορών που θα στηρίζονται στον κίνδυνο που ενέκρινε το προηγούμενο, προηγούμενο κοινοβούλιο και ε, αν έχουμε εξάντε προσδιορισμένες συνεισφορές ως πάγιο ποσοστό των καταθέσεων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το προφίλ του κινδύνου, είναι σαφές ότι τα ιδρύματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε ηθικό κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των συνεισφορών στο σύστημα εγγύης καταθέσεων, η ομάδα μας θέλει το άρθρο, να διατηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 13. Δηλαδή το σύστημα εγγύης καταθέσεων, το DGS, να αναπτύσσεται και να χρησιμοποιεί τις δικές του μεθόδους υπολογισμού για να ε, προσαρμόσει τις συνεισφορές ε, στα προφίλ κινδύνου και στις κατάστασεις της αγοράς. Επίσης, ε, μπορεί, μπορούν τα κράτη-μέλη για κλάδους χαμηλού κινδύνου και για συγκεκριμένα μέλη e IPS να προβλέπουν τα κράτη-μέλη χαμηλότερες συνεισφορές. Ε, βέβαια, ο σκιώδη Ηγητής ακόμη εξετάζει τι κατευθυντήριε γραμμές, ε, αλλά ήδη εντόπισε μερικά θετικά του σημεία. Οι αρμόδιες αρχές ε, μπορούν να αποκλείσουν ένα ε, ίδρυμα, την εξαίρεση ενός κινδύνου για ένα ίδρυμα, εφόσον ο δείκτη αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι διαθέσιμος. Και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προβλέψουν επιπλέον δείκτες κινδύνου αν θεωρούν ότι οι βασικοί δείκτες δεν λαμβάνονται όντως υπόψη τα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων μελών. Για παράδειγμα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη ενός IPS ή ε, να καλυφθούν κάποιοι κλάδοι με χαμηλό κίνδυνο που εμπίπτουν στο στην εθνική νομοθεσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μέθοδο ε, αξιολόγηση, ίδια μέθοδο αξιολόγηση κινδύνου και εδώ θα πρέπει να τηρηθούν οι κατευθυντήριε γραμμέ ε, όταν εφαρμόζονται οι ίδιε μέθοδοι για τον κίνδυνο για τον υπολογισμό του κινδύνου. Σε ό,τι αφορά τι υπόλοιπε κατευθυντήριε γραμμέ, ε, θα θέλαμε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν οι σκιώδει ηγητέ να έχουν εκτενεί διαβουλεύσει στι πολιτικέ ομάδε πριν αποκρισταλώσουν τη γνώμη του. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Τέρχο. Δεν βλέπω κανέναν του φιλελευθέρου. Τι καλά, ούτε γκου έχουμε. Αγαπητέ κύριε Σβέν Γκίγκολτ, έχει το λόγο εσύ. Αγαπητέ Μάρκο. Βλέπουμε εδώ από τη θέση που κάθομαι αν είναι κανείς παρόν ή όχι. στο πνεύμα της δημοκρατίας είναι αυτό το να μπορούμε να παρακολουθούμε ποιος είναι παρόν και ας μιλήσω αγγλικά καλύτερα. Πέραν των ερωτημάτων που εγείρουν οι συνάδελφοι εδώ και με τα οποία συμφωνώ, έχω μία ερώτηση η οποία είναι γενικότερο ενδιαφέροντος. Το EPA όταν αποφασίσαμε εμείς για τον κανονισμό του είχε σαν ξεκάθαρη εντολή να υποστηρίξει την αναλογικότητα Υπήρξε και μια ομάδα εργασίας πριν ένα χρόνο. Πολλοί συμμετείχαν εκεί, έγιναν πολλές συζητήσεις. Από τότε όμως δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Μπορείτε να μας πείτε τι συγκεκριμένα μέτρα έχετε πάρει έτσι ώστε να στηριχθεί αναλογικότητα. Και το νέο κύμα αυτό των ρυθμίσεων δεν δημιουργεί προβλήματα στους μικρότερους εταίρους ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους και το, τα κέρδη τους κινδυνεύουν να πληρώνουν περισσότερα. Θα μπορούσε λοιπόν το IPA να μπορέσει να πει στο Κοινοβούλιο τι μέτρα έχουν ληφθεί στον τομέα της αναλογικότητας και σε ποιο βαθμό ε, θα ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα εργασίας για τη βελτίωση της κατάστασης, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχετε αγνοήσει την προοπτική αυτή της εντολής την οποία σας έχει δώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα, έρθω με την, θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Εγώ δεν είπα ότι η EBA θα ε, ε, μπορεί να δώσει περισσότερα στοιχεία στην παρούσα φάση, αλλά θα μεταφέρω την ερώτησή σας και θα επανέλθουμε γραπτά. Πάντως μπορώ να απαντήσω επί της ουσίας. Εγώ ίδιος τους τελευταίους μήνες λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας το θέμα της αναλογικότητας με διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι εδώ αντιστοιχούμε τις προσπάθειές μας με το επίπεδο της ευελιξίας. Ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση και σε σχέση με τη διαχείριση των εγγυήσεων που είναι διαθέσιμες, δηλαδή να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Είχα εδώ ένα παράδειγμα αλλά δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Να επανέλθω η ευελιξία γενικότερα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ και δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι μαγικό. Το επιχείρημα παρουσιάζεται και από την άλλη πλευρά. Ακόμα και με το 100% της εξίσωσης εναρμονισμένο. Εφόσον δεν εναρμονίζουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονται οι δείκτες, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Να σας πω γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να εναρμονίσουμε μερικά πράγματα. Παίρνετε το επίπεδο κεφαλαίου σαν παράδειγμα και αποφασίζετε ότι θα, ε, ότι θα συνδέσετε διάφορες ταθμίσεις πάνω σε αυτό. Η κοινότητα των πιστοτικών ιδρυμάτων βέβαια σε κάθε χώρα διαφέρει από μια άλλη χώρα έτσι ώστε αν δώσετε ε, ένα ανώτατο όριο για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στη μία χώρα και στην άλλη χώρα. Δεν υπάρχει μια αντίστοιχη ε, θα έλεγα παρουσίαση. Μου είπατε αν το 25% είναι ικανό ποσοστό ευελιξίας ενώ το 75% είναι ένα αρμονισμένο ποσοστό. Το θέμα είναι σε όλα αυτά τα ποσοστά και κυρίως το 75% να υπάρχει μια εσωτερική ευελιξία. Σχετικά με τον εντολή όπως είπε ο κύριος Γκίλγκοντ. Εμείς προωθούμε στα πλαίσια της εντολής την σύγκληση στις πρακτικές εποπτείας και ελέγχου. Ακούγεται περίπλοκο αλλά δεν είναι θα ήταν λάθος ε, να προωθήσουμε εμείς ε, ε, κάποια εναρμονισμένα πλαίσια αν δεν δώσουμε πιο συγκεκριμένες οδηγίες και στοιχεία. Τώρα για το IPS. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ και υπάρχει μια κάποια σύγχυση. Υπάρχουν τα μέλη τράπεζες σε ένα IPS και ταυτόχρονα και σε ένα επίσημα αναγνωρισμένο DGS. Το θέμα είναι ότι έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα επειδή είναι μέλη του IPS και όταν έρχονται ε, στα πλαίσια των επίσημα αναγνωρισμένων DGS τότε υπάρχει αναγνώριση της ε, ε, αυξημένης αντοχής τους μέσω της επιβολής μικρότερης συμμετοχής. Δεν είμαστε στο 1% ακόμα, κατά λάθο το είπα, είμαστε στο 0,8%. Λοιπόν, όλες οι τράπεζες που είναι σε IPS και σε DGS ε, δεν είναι ε, ε, εκτός κινδύνου πλήρως, οπότε δεν μπορεί σε όλες αυτές τις τράπεζες να επιβάλλει κανείς μικρότερο ποσοστό επιβολής. Και εδώ έρχομαι σε αυτά που είπε και ο κύριος Μπάλτς και ο κύριος Σιμών. Ο ενδογενής κίνδυνος είναι κάτι το οποίο ξεπερνά ε, τη βάση των καταθέσεών τους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν ε, τα κεφάλαια των τραπεζών αυτών και θα πρέπει να υπερασπιστούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι τώρα. Εφαρμόζουμε με εξαντλητικό τρόπο το 13-2. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή να μην λάβουμε υπόψη μας στο επίπεδο των καταθέσεων. Όχι το σημείο εκκίνησης είναι η κάλυψη των, ε, των ε, καταθέσεων. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να το αγνοήσουμε αυτό και ε, να μην αγνοήσουμε την εξωτερική επιπλέον διάσταση την οποία αποκτούν μέσω της συμμετοχής τους στις εξωτερικές αυτές οντότητες. Σας ευχαριστώ. Εισηγητής. Αν δεν υπάρχει κανείς άλλος. Πέτσερ. Ευχαριστώ πολύ. Μα ακριβώς εδώ θέλω να απαντήσω. Δεν είναι το θέμα η προσαρμογή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ πιο βασικό. Δηλαδή να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε ορίσει στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Μια μέθοδο στηριγμένη στον ίδιο κίνδυνο με τις συνεισφορές αναλογικά του επίπεδου κινδύνου των μελών. Όλα τα συστήματα ε, διασφάλισης καταθέσεων, όπως και να τα πείτε δεν με νοιάζει, είναι τελικά ισότιμα. Δεν, δεν θα πούμε ότι ένας πληρώνει περισσότερο ή λιγότερο, αλλά μέσα στο σύστημα αυτό πρέπει αυτός που έχει μεγάλο κίνδυνο να πληρώνει. Δηλαδή οι πιο τα πιο κεντρικά ιδρύματα. Εκεί πέρα έχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Έτσι λοιπόν, στην, ε, στον επιμερισμό του κινδύνου μπορούμε να έχουμε την ίδια αναλογία όπως έχουμε τώρα. Τα όρια δηλαδή τα οποία χαράστε εσείς είναι τα μαθηματικά όρια. Με τα μαθηματικά όρια εκείνος που έχει μεγαλύτερο κίνδυνο στο μέλλον θα πληρώνει λιγότερο. Αυτό δεν, το δέχομαι λοιπόν. Το λέω ξεκάθαρα. Και από αυτή τη θέση. Είμαι διαμετρικά αντίθε... είναι διαμετρικά αντίθετο αυτό που λέτε προς αυτό το, το οποίο εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε ζητήσει με την νομοθεσία. Δηλαδή, κίνδυνο αναλογικό και εισφορά αναλογική του κινδύνου. Αυτός που έχει υψηλό κίνδυνο θα δώσει περισσότερο χρήμα γιατί διαφορετικά θα πρέπει να καλυφθεί από το χρήμα του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Και αυτό θα σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν θα αναλαμβάνει κίνδυνο ελαφρά την καρδία, αλλά θα αναλογίζεται ότι σιγά σιγά αυτός ο κίνδυνος του καθίσταται και πιο ακριβώς. Και πρέπει και αυτό να το λάβει υπόψη. Έτσι λοιπόν, αυτά τα συστήματα διασφάλισης πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν και στο μέλλον όπως λέει και ο κανονισμό, στο άρθρο 26, ο κανονισμό της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής, άρθρο 26 λοιπόν, ότι πρέπει τα συστήματα διασφάλισης να λειτουργούν απρόσκοπτα, γιατί όπως το έχετε τώρα, θέτουμε ε, σε κίνδυνο και αυτά τα συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος συνάδελφος θέλει ενδεχομένω να λάβει το λόγο. Όχι. Κύριε Κανόνα. Ε, <clears throat> yes. Again, I... Ευχαριστώ. Ίσως, ίσως να μην τα διευκρίνησα καλά. Αναφέρεστε στα στοιχεία όπως έχουν δημοσιευθεί. Στο 25% υπάρχει μια εσωτερική ρύθμιση λοιπόν, η οποία αυτή όμως δεν αρκετεί. Γι' αυτό το εξετάζουμε το θέμα. Συμφωνούμε μαζί σας λοιπόν σε αυτό. Αν το εισάγουμε αυτό σαν παράμετρο της ελάχιστης συνεισφοράς είναι ένα συν, δεν είναι πολλαπλασιαστής, οπότε έχετε ένα περιθώριο αξιολόγησης πολύ ευρύτερο. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε άλλο τρόπο για να δείξουμε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ που ήρθατε από το Λονδίνο κύριε Κανόνα για να μιλήσετε στην Επιτροπή μας. Αν βλέπω σωστά στην ημερήσια διάταξη, δεν έχουμε τίποτα άλλο για σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ και θα σας ξαναδώ ελπίζω στις 3 το απόγευμα μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής των Εσωτερικών για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της οδηγίας για την νομοποίηση παρανόμων εσόδων. Πέρα στην μεριά σας.